παρακαλώ αναφερθείτε στο θέμα της διαδικασίας. Είναι νομικό θέμα που συνέβη στην χώρα μου, που θεωρώ πως αφορά το σώμα. Απαλλάχθηκα από όλες τις κατηγορίες ε, ε, που υπήρχαν εναντίον μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που με στήριξαν. Από όλες τις πτέρυγες είχα στήριξη από πολλούς συναδέλφους από πολλές χώρες και μου είπατε καλό κουράγιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο εδώ πέρα, τον Άγνιου, τον ε, Πολ Νάτα, τον Νάιτζελ Φάρατζ που ήταν σε επαφή, τους συναδέλφους από το ENF. Εσείς πιστέψατε σε μένα. Θα ήθελα να ξεχωρίσω τρία άτομα. Τον Έντουαρτ Φαράντ, πάρα πολύ καλή ε, πολιτικό, και την Μαρίν Λεπέν, την οποία ευχαριστώ. Οι ευχαριστίες σας δεν είναι επί της διαδικασίας. Σας παρακαλώ να μην καταχράσετε τις ανεκτικότητες του προεδρίου και να μην παραβιάζετε τον κανονισμό. Μπορούσατε να του στείλετε λουλούδια και όχι αυτή τη στιγμή. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Έχουμε την έκθεση Χάουταλα ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Λαβία. Ψηφοφορία επίσης με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε επίσης στην επόμενη έκθεση Λαβία, επίσης με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Κάουφμαν, Επίσης, ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Γκρίσμπεκ. Επίσης με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Χρυσόγονου για την αίτηση άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Γιάτσεβιτς. Ψηφοφορία με ανάταση της χειρός. Πώς είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη έκθεση επίσης του κυρίου Χρυσόγονου, αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του ίδιου συναδέλφου για άλλο θέμα, με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Φεράρα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Φιλιππό με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε Πυρίνσκη. Υπάρχει η τροπολογία 62 με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά συνέπεια περνάμε τώρα στην τροπολογία 64 ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62 με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 63 ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται η πρόταση της επιτροπής ψηφοφορία με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το νομοθετικό ψήφισμα ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Demesmaeker. Εδώ θα έχουμε περισσότερες ψηφοφορίες. Στην παράγραφο 11 σε τρία μέρη με ανάταση της χειρός. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος υπέρ να κάνουμε εφόσον το ζητάτε παρότι ήταν καθαρό το αποτέλεσμα έλεγχο στο δεύτερο μέρος της παραγράφου 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Ε, το τρίτο μέρος της παραγράφου 11 με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 29 με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 31 σε δύο μέρη με ανάταση της χειρός. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 40 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 41 με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 42. Με ανάταση της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 58 σε τρία μέρη. Είναι σαφής η πλειοψηφία, συνάδελφοι, μην επιμένετε. Ε, σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές να κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο μέρος της παραγράφου 58. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία ελπίζω να μην ξαναζητήσετε τσεκ να σέβεστε το προεδρείο και την κρίση του. τρίτο μέρος με ανάταση χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 72 με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 78 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ... No, uh, Συγγνώμη, επαναλαμβάνουμε στην παράγραφο 71 παράγραφος 71 το αρχικό κείμενο σε τρία μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 72 το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 78 σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές σε αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε έλεγχο. Παρακαλώ με το δεύτερο μέρος της παράγραφου, της παραγράφου 78 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε με μικρή διαφορά. Παράγραφος 80 σε δύο μέρη. Το πρώτο τμήμα με ονομαστική με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος παραγράφου 80 ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, υπάρχει μια τροπολογία, η τροπολογία 2 μετά την παράγραφο 80 με ανάταση της χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 81 σε δύο μέρη με ονομαστική κλίση το πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται δεύτερο μέρος της παραγράφου 81 με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 82 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 88 επίσης με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίνεται. Τροπολογία 3 μετά την παράγραφο 90 με ανάταση της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με ανάταση της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφοφορία στο σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούν οι επεξηγήσεις ψήφου.